Meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που έχουμε μαζί μας σήμερα τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Γεωργίας, τον κύριο Ούζου Πασφίλη. Σας καλωσορίζω λοιπόν ε, στην Επιτροπή μας σήμερα. Νομίζω ότι έρχεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονική συγκυρία. Βρισκόμαστε στη φάση προετοιμασίας της Σύνοδου του Vilnius. Το πολιτικό σενάριο στην Γεωργία τροποποιείται, μεταβάλλεται. Για πρώτη φορά καταφέραμε σε μία από τις χώρες αυτές να γίνει μία ειρηνική μετάβαση σε μία άλλη α, ε, μορφή εξουσίας και θέλουμε φυσικά να υπάρχει δυνατότητα τέτοια ειρηνική αλλαγή της ε, εξουσίας γιατί αυτό εκφράζει πραγματικά η ύπαρξη δημοκρατίας και κράτος δικαίου ότι υπάρχουν οι απαραίτητοι όροι και ότι συνεχίζουν να εξελίσσονται προκειμένου να υπάρχει τέτοια δυνατότητα και βλέπουμε ότι οι διαπραγματεύσεις για την Συμφωνία Εταιρική σχέση ε, προχωρούν. Θα δούμε κατά πόσον θα καταφέρουμε να ολοκληρωθούν. Θεωρούμε από πλευρά μα ότι είναι σημαντική χώρα η Γεωργία, μια σημαντική χώρα, λέγω, από μόνη της, αλλά και λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε οι μελλοντικές εξελίξεις να, μας, να συνδέσουν τη χώρα αυτή με την ευρωπαϊκή προοπτική, αλλά και με τις ευρωπαϊκές ε, αξίες της ε, δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Κύριε Πρόεδρε, θα ήμουν ευγνώμων αν μου δίνετε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε, σχέσεις, να αλλάξουμε ε, απόψεις για την εξέλιξη της χώρας σας και της δημοκρατίας στη χώρα σας. Έχετε το λόγο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για το χρόνο που αφιερώνετε στη χώρα μου, στη Γεωργία και σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να παραβρεθώ ενώπιόν σας και να απαντήσω στις ερωτήσεις που ενδεχομένω έχετε για τις πρόσφατες εξέλιξεις στη Γεωργία. Τα τελευταία 23 χρόνια όταν ε, η γεωργία ε, θεωρούταν ε, κατά της Ευρώπης η υποστήριξή σας ε, στη χώρα μου ήταν ουσιαστική και σας ευχαριστώ. Ακόμη και τώρα το γεγονός ότι ζούμε σε ένα πάνω κάτω ειρηνικό περιβάλλον αλλά το ότι ένα μεγάλο μέρος της επιτράτειας της Γεωργίας είναι η παροσική κατοχή ακόμη Ναι, επειδή η αποστολή παρακολούθησης της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στη Γεωργία και αποτρέπει την επιδείνωση της κατάστασης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή που προσδίδετε στη χώρα μου και στην προθυμία σας ε, να βρεθούν τρόποι για να γίνει ακόμη πιο στενή και αποτελεσματική η συνεργασία. Και πριν από τη Σύνοδο Κορφής ε, του Βίνιους, το ότι θέλετε να συζητήσουμε τις πρόσφατες εξελίξεις δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη βούληση να μας βοηθήσετε σε αυτή τη διαπραγματευτική διαδικασία και να αυτή η διαδικασία με επιτυχία. Έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές αυτόν τον Νίκο, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Στο παρελθόν ερχόμουν εδώ ως ένας από τους ηγέτες της ε, αντιπολίτευσης ή ένας από τους επικεφαλείς της κοινωνίας ε, των πολιτών. Και ε, ξέρετε, είναι δύσκολο να έχει κάποιος το άχθος της διακυβέρνησης. Η νέα κυβέρνηση ανέλαβε επικεφαλής της από τα τέλη Οκτωβρίου 2012 και ναι, από Είδαμε ότι από τις εκλογές και μετά είχαμε πάρα πολύ σημαντικά πολιτικά μηνύματα για τη χώρα μου. Ήταν η πρώτη φορά οι εκλογές ε, αποτέλεσαν το φόρουμ της αλλαγής. Και φυσικά αυτό είναι κρίμα για μια χώρα που είναι ανεξάρτητη εδώ και 22 χρόνια και δεν ε, κατάφερε να έχει νωρίτερα αυτή την εξέλιξη. Όμως ε, τελικά συνέβη και θέλουμε να οικοδομήσουμε από αυτό. Πρόεδρε, εγώ ακολουθώ τη συμβολή για απαραίτητες αλλαγές στο μέλλον. Όταν ε, οι εκλογές θα πρέπει να καταλήξουν στο να έρθουν νέοι άνθρωποι στην εξουσία. Είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η συμβουλή και το μήνυμα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το κύριο ζήτημα αυτής της συμφωνίας ε, μεταξύ μου και των προηγούμενων ε, κυβερνητικών αρχηγών και του Προέδρου Σασκασβίλη είναι αμέσω μετά την επαναστασία και το δικό μου κόμμα και κάποιοι άλλοι ε, αγωνιστήκαμε για να νικήσουμε την προηγούμενη κυβέρνηση και του είπαμε ότι το πρώτο θέμα στην ατζέντα του δημοκρατισμού της χώρας θα πρέπει να είναι πώς θα πορευτούμε μετά τις εκλογές, πώς θα διακυβερνήσουμε. Βέβαια δεν ακούστηκε το μήνυμα αυτό, δυστυχώς, και όλα αποσκοπούσαν ε, στο να διατηρηθεί ένα μονολυθικό σύστημα εξουσίας που τελικά άλλαξε με την νέα κυβέρνηση. Κατά τους τελευταίους 7-8 μήνες είχαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο γιατί για πολλά χρόνια μας αποκαλούσαν την αντιπολίτευση του δρόμου, γιατί δεν υπήρχε κανένας χώρος για την αντιπολίτευση στο κοινοβούλιο ή στα τοπικά συμβούλια, φυσικά στην κυβέρνηση. Και επομένω υπήρχαν κάποιε ανησυχίε. Ποιο ήρθε στην εξουσία. Είναι πολύ δύσκολο να πιστέψει κανεί ότι στη Γεωργία για πολλά χρόνια αυτοί που κυβερνούσαν τη χώρα και έδειχναν τάσεις υπέρ της, και θέσεις υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ του ΝΑΤΟ και για την αντιπολίτευση το απλό συμπέρασμα ήταν ότι αυτοί μάλλον θα είναι φιλορώσοι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά του ΝΑΤΟ. Έτσι λοιπόν φαινόταν σαν να παραγόνται δύο είδη πολιτικών ηγετών και τάσεων και πιθανότητα κατά τους τελευταίους 6-7 μήνες εμείς αποδείξαμε ότι ο πολιτικός συνασπισμός στο γεωργικό όνειρο όπου συμμετέχουν ε, και 6-7 κόμματα και το κόμμα του οποίου πρόεδρος είμαι εγώ, μέλος ε, της ε, Διεθνού των φιλελευθέρων. Έχουμε λοιπόν τη συμμετοχή αυτού του κόμματο, τη συμμετοχή του συντηρητικού κόμματο, όχι σχέση με το ECR. Έχουμε το νέο κόμμα που ιδρύθηκε από τον κύριο Βενσβίλη, το Γεωργιανό Όνειρο, όπως αποκαλείται και ο συνασπισμός, και έχουμε και το ε, Εθνικό Φόρουμ, έχουμε το ε, βιομηχανικό κόμμα. Έτσι λοιπόν ε, είναι ευρία η συμμετοχή στο συνοφισμό, έτσι όμως κατορθώσαμε να αποδείξουμε ότι η στρατηγική για τη Γεωργία δεν αλλάζει. Η καλύτερη αποδείξη ήταν το ψήφισμα του Κοινοβουλίου το Μάρτιο προετοιμάστηκε και ψηφίστηκε και από την πλειοψηφία και τη μειοψηφία και υιοθετήθηκε από κοινού και σε αυτό το έγγραφο και πάλι υπογραμμίζονται οι στρατηγικοί μας στόχοι. Καταστήσαμε σαφές ότι η Ευρώπη είναι ο μόνος προορισμός που μπορούμε να σκεφτούμε και ότι η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και ένταξη στο ΝΑΤΟ, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ είναι μονόδρομος. Ε, δεν σκεφτόμαστε κάτι άλλο, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική για να είναι ασφαλής και ευημερής και ειρηνική η χώρα μας. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου ακολουθεί νέες προσεγγίσεις η νέα κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί το κύριο πρόβλημα με τη Ρωσία. Στο έγγραφο υπογραμμίζουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει και τίποτα δεν θα γίνει το οποίο θα αμφισβητήσει την ένταξή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και αν οτιδήποτε αντίκειται σε αυτή τη στρατηγική επιλογή, δεν μας αφορά και ταυτόχρονα ακούμε πάρα πολύ σοβαρά τις συμβουλές από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ ότι πρέπει να βάλουμε την δυνατά μας για να εξομαλύνουμε τις σχέσεις με τη Ρωσία. Αρχίσαμε λοιπόν να εντοπίζουμε κάποια θέματα χαμηλού προφίλ για να αρχίσουμε τις επαφές ε, και ο Πρωθυπουργό έχει υλοποιήσει τρει γύρου συναντήσεων για τη σχέση με τη Ρωσία. Συζητάτε πώ η Ρωσία θέλει να εφαρμόσει τι υποχρεώσει της για την προσχώρηση στον ΠΟΕ όταν έγινε αυτό και να ανοίξει τις αγορές για τα προϊόντα της Γεωργίας. Πώς να διασφαλιστεί ότι οι Γεωργιανοί πολίτες ε, που ζουν στη Ρωσία, το 15% του πληθυσμού ζει στη Ρωσία, μπορούν να έλθουν στη Γεωργία, να επισκεφτούν τις οικογένειές τους και τους συγγενείς τους. Επίσης, θέλουμε να συζητήσουμε το θέμα των μεταφορών και των συνδέσεων. Γιατί ξέρετε, από το 2008 ακυρώθηκαν οι ε, μεταξύ Μόσχας και Τυφλίδα. Έτσι, λοιπόν, θέλουμε να βρούμε λύσεις σε αυτά ε, και στα θέματα που φέρνουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε θέματα τελωνιακής ένωσης, σε θέματα ασφαλείας. Ε, αυτά δεν είναι αποδεκτά από εμάς έτσι όπως τα προτείνουν οι Ρώσοι. Για διαπραγματευτικέ διαδικασίες τώρα πριν από τη σύνοδο στο Βίλνιους προοδεύουν καλά και σήμερα συνεχίζονται οι συζητήσεις για το θέμα αυτό και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να υπογράψουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης με όλα σε επιθυμούμε, με τα απαραίτητα χαρακτηριστικά. Επίση, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να εργαστούμε και εμεί από την πλευρά μα για να αποδείξουμε σε όλου ότι έχει νόημα συνεργασία με τη Γεωργία και ότι μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι εταίροι. Παραδείγματο χάρη, ο εργατικό κώδικα, που για χρόνια αποτελούσε αντικείμενο διένεξη μεταξύ τη κυβέρνηση και διεθνών οργανισμών και όχι μόνο του ΔΕΛΑ και το αμφισβητούσε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κοινοβούλιο έκανε μια εντατική δουλειά πολύ δύσκολη δουλειά το τελευταίο εξάμεινο και υιοθετήσαμε τροποποιήσεις στον εργατικό κώδικα που είναι τώρα αποδεκτές από το Διεθνή Οργάνωση Εργασία, από τις πολιτικές δυνάμεις, από τους εμπειρογνώμονες, από τα συνδικάτα και πιστεύουμε ότι έτσι θα βελτιωθούν τα πρότυπα της νομοθεσίας και να προσεγγίσουμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Κυρώσαμε τα έγγραφα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και πριν δύο εβδομάδες ένας, ε, διορίστηκε ένας ειδικό επιθεωρητής για την προστασία των δεδομένων, επιλέχθηκε από την κοινότητα των ΜΚΟ και είχε και την απαραίτητη εμπειρία για το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα δυστυχώς, γιατί οι νέοι επικεφαλής της αστυνομίας ανακάλυψαν στα αρχεία της αστυνομίας εκατοντάδες παράνομες κασέτες που για πολλά χρόνια ηχογραφούνταν και παρακολουθούνταν ιδιωτική ζωή πάρα πολλών ανθρώπων, όχι μόνο πολιτικών της αντιπολίτευσης. Και αυτά τα αρχεία έχουν για προφανείς λόγους. Βέβαια αποφασίστηκε ότι θα καταστραφούν αυτά τα αρχεία και θα παρευρίσκονται και ειδικοί εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών για να επαληθεύσουν την καταστροφή και για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Ο Υφυπουργό Ιστορικών που διορίστηκε πριν ε, λίγους μήνες ε, συνελήφθη και αποπέμφθηκε γιατί αποκαλύφθηκε ότι συνδεόταν με αυτά τα θέματα. Επίσης, έχουμε ξεκινήσει σημαντική μεταρρύθμιση στο δικαστικό σύστημα. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας έχουν οι δικαστές το δικαίωμα να ε, κλέξουν ε, τους εκπροσώπους τους ε, στο ανώτατο δικαστήριο. Είχαμε εκλογέ ο κάθε δικαστής μπορούσε να καταθέσει την υποψηφιότητά του στο παρελθόν ο επικεφαλής ε, των δικαστών ε, είχε το δικαίωμα να διορίζει τους υπόλοιπους δικαστές, ενώ σήμερα βλέπουμε ότι το σύστημα πραγματικά αποτελεί, ε, αποκτά πραγματική ανεξαρτησία από τους πολιτικούς θεσμούς. Επίσης, ε, προετοιμάζεται και ένα νομοσχέδιο. Έχουμε ανταλλάξει εμπειρίε με χώρε τη Ανατολική Ευρώπη από την Πολωνία. Οι εμπειρογνώμονε μα ε, επισκέπτονται την Πολωνία και πρόκειται να ε, θεσπίσουμε ένα αποκεντρωμένο σύστημα διακυβέρνηση. Μέχρι τώρα είχαμε ένα συγκεντρωτικό σύστημα διακυβέρνηση, το οποίο ήταν αποτελεσματικό για την επιτύχηση ορισμένων στόχων, αλλά δεν ήταν αποτελεσματικό για να καταστούν οι άνθρωποι ανεξάρτητοι και υπεύθυνοι στη ζωή του. Αρχίσαμε μεταρρυθμίσεις ε, στη μεταναστευτική πολιτική και στη σχετική υποδομή θα έρθει σε δύο εβδομάδες ε, το νομοσχέδιο στο Κοινοβούλιο και λαμβάνουμε αυτό το θέμα πάρα πολύ σοβαρά. Κυρίω μετά την πρόοδο που σημειώθηκε με το θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Μέχρι τώρα η Ρωσία ήταν υπερβολικά ελεύθερη προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, έχει ε, ένα καθεστώς ε, διευκόλυνσης ε, θεώρησης με πάνω από 200 χώρες στον κόσμο, η Γεωργία, αλλά βέβαια θα πρέπει να αλλάξει η πολιτική μας ε, σε αυτό το θέμα. Το θέμα των μειονοτήτων είναι κρίσιμο, είναι ζωτικό για τις νέες δημοκρατίες. Ο νόμος για την απαγόρευση εισαγωγής διακρίσεων θα έρθει στο Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο λαμβάνονται συγκεκριμένα βήματα και είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός της χώρας ακολουθεί αυστηρή πολιτική για το θέμα αυτό και στις δηλώσεις του καθιστά σαφές πως οποιαδήποτε αιτιολόγηση για οποιαδήποτε εισαγωγή διάκρισης κατά των μειονοτήτων, είτε είναι θρησκευτική πολιτικές μειονότητες, γλωσσικές μειονότητες λοιπά Δεν θα το ανεχτούμε αυτό. Γιατί, ξέρετε, στο Κεφτεμέου πάρα πολλοί συνελήφθησαν και συνεχίζονται οι έρευνες και κατά δύο εκπροσώπων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας, οι οποίοι είχαν ε, κάνει κάποιες παράνομες πράξεις. Τώρα συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. Κατά το τελευταίο ένα μήνα δυστυχώς χάσαμε 10 στρατιώτες. Ε, αυτό είναι το 1 τρίτο των συνολικών θυμάτων της Γεωργίας μας σε ε, τρία χρόνια, παρουσίας μας εκεί. Αλλά ξεκαθαρίσαμε σε όλους ότι δεν θα υποχωρήσουμε λόγω αυτού παρά το ότι υπάρχουν κάποιες εκκλήσεις από τον κόσμο. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν ερωτήσεις γιατί είμαστε εκεί, γιατί έχουμε παρουσία εκεί, όμως η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι δεν θα υποχωρήσουμε. Το αντίθετο μάλιστα δεσμευτήκαμε ότι θα υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορες αποστολές ε, και στο Μάλι. Και οι στρατιώτες μας είναι έτοιμοι να συμμετέχουν στην αποστολή. Εμείς προσπαθούμε να συνεχίσουμε τις επιτυχίες της προηγούμενης κυβέρνησης εκεί όπου είχε σημειωθεί επιτυχία, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να αλλάξουμε και όσα δεν είχαν γίνει σωστά. Επομένως, έχουμε ιδιαίτερες προκλήσεις μπροστά μας, υπάρχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες από τους πολίτες, γιατί κληρονομήσαμε μια χώρα που πάνω από το 50% του πληθυσμού πιστεύει ότι είναι άνεργη και το 45% των οικογενειών έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα παροχής κοινωνικής βοήθειας. γιατί ζουν ε, κάτω από το όριο της φτώχειας. Έτσι λοιπόν, δυστυχώς οι επιτυχίες που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια δεν οδήγησαν στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών στη χώρα μας και εμείς πρέπει να εργαστούμε πολύ σκληρά. Και πάλι, σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας, για την προσοχή σας, για την ετοιμότητά σας να λάβετε σοβαρά υπόψη τη Γεωργία και σας ευχαριστώ και για τις συστάσεις και για τις ερωτήσεις σας, τις εκτιμούμε ιδιαίτερα. Και πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και στα τέλη του έτους θα μπορέσουμε να πούμε ότι η Γεωργία βρίσκεται σε ένα ακόμη ψηλότερο επίπεδο ολοκλήρωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, ότι θα αυξηθούν και οι ευκαιρίες που αναμένουμε από αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ανοίξουμε λοιπόν τώρα τη συζήτηση. Ο κύριος Λίζακ είναι ο πρώτος ομιλητής, ο οποίος είναι και εισηγητής για τη Γεωργία. Ευχαριστώ Πρόεδρε να μιλήσω στα πολωνικά. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω και να σας καλωσορίσω. Βρισκόμαστε κάθε κάποιες εβδομάδες, νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα καλό σημάδι. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα Στη σημερινή όμως ε, κατάσταση θα πρέπει να σας πούμε ότι ο κύριος Μασισβάλλη, ο πρώην ε, πρωθυπουργός, ξεκίνησε απεργία πείνας σήμερα. Και αυτό έχει να κάνει με την απαγόρευση που του επιβλήθηκε να επανανεωθεί με την οικογένειά του. Επίσης δεν έχει πρόσβαση στην τηλεόραση, σύμφωνα με την γεωργικό νόμο θα έπρεπε να έχει τέτοιες δυνατότητε. Όπως αναφέρθηκε και εξ αρχής, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερως για το γεγονός ότι η συνεργασία σας με την αντιπολίτευση στο Κοινοβούλιο διατηρείται σε επίπεδα που αρμόζουν σε μία δημοκρατία. Γνωρίζουμε από τον κύριο Μπακράζα, εκπρόσωπο της αντιπολίτευση, ότι η συνεργασία είναι καλή. Φυσικά, τα πράγματα δεν είναι απλά, υπάρχουν πολιτικές εντάσεις, πολιτικές τριβές, παρόλα αυτά η συνεργασία αυτή είναι πολύ καλή. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό είναι ένα σημάδι επικοδομητικής πραγματικά διάθεσης και συνεργασίας από πλευράς του κόμματος της κυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης. Θεωρώ ότι είναι μια κατεύθυνση την οποία υποστηρίζουμε. Για τα ιστορικά ζητήματα τώρα τα οποία αναφέρατε θα ήθελα να πω το εξή. Ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργό στην τελευταία επίσκεψη στη Γεωργία δεν έκρυψαν ότι η κατάσταση πραγματικά είναι τεταμένη. Αυτό μη θεωρήσετε παρακαλώ ότι αποτελεί προσωπική επίκριση εδώ. Ε, Αντιπροσωπεύετε και τον κυβερνητικό συνασπισμό, όχι μόνο το δικό σας κόμμα και τον εαυτό σας ασφαλώς. Ως εκ τούτου θα ήθελα να σας παρακαλέσω και να σας θέσω το εξής ερώτημα. Πώς θεωρείτε εσείς ως κυβερνητικός ε, συνασπισμός, πώς αξιολογείτε το μοντέλο ε, λειτουργίας της δημοκρατίας. Πώς θέλετε ότι λειτουργεί η δημοκρατία και πώς θα έπρεπε να λειτουργεί η δημοκρατία σας. Εμείς να σας πούμε ότι απ' έξω, παρά το γεγονός ότι δεν ε, βλέπετε σε τη σύγκριση αυτή, εμείς αναρωτιόμαστε κατά πόσον η κατάσταση στην Γεωργία ε, προσωμιάζει αυτή της ε, Ουκρανίας. Η πρώην Πρωθυπουργός του Μοσέγκο έχει συλληφθεί και κατηγορείται Όπω και κατηγορείται και ο πρώην Πρωθυπουργός Μενετσίλη. Είναι λοιπόν παρόμοια η κατάσταση, ασφαλώς και υπάρχουν διαφορές. Η κυρία Τιμοσέγκο. Κρατείται σε μια πολύ καλύτερη φυλακή. Έχει πρόσβαση τουλάχιστον στην τηλεόραση, σε ενημέρωση. Και γι' αυτό λοιπόν ρωτώ Πώς θεωρείτε λοιπόν θα εξελιχθεί στο μέλλον η συνεργασία της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Σουπασπέλη. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την Γεωργία για την ειρηνική αυτή μετάβαση. Έγιναν αλλαγές στην κυβέρνηση χωρίς δυσκολίες, χωρίς ε, να Η Γεωργία μέχρι τις τελευταίες εκλογές ήταν μια χώρα με ένα κόμμα, μονοκομματική, με αυταρχική ηγεσία. Δεν υπήρχε αντιπολίτευση, δεν υπήρχε αντιπολίτευση στο κοινοβούλιο, δεν υπήρχε συνεργασία με κανέναν από την αντιπολίτευση. Χαίρομαι λοιπόν που ο κύριος Λίσεκ τώρα ζητάει συνεργασία ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Γιατί ακριβώς αυτό είναι που έλειπε από τη Γεωργία. Αυτό ακριβώς είναι που χρειάζεται η Γεωργία. Βρίσκεται σε μετάβαση από το μοναδικό σύστημα στο πολυκομματικό σύστημα η Γεωργία. Άρα πρέπει να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις ειρηνικά. Τα κόμματα που είναι στην κυβέρνηση πρέπει να αποφύγουν αδυναμίες, σφάλματα που έχουν διαπράξει οι προηγούμενοι κυβερνώντες. Μια παγίδα στην οποία θα μπορούσε να πέσει η κυβέρνηση θα ήταν μια πολιτική βεντέντα. Ξέρουμε ότι η κοινωνία της Γεωργίας πιέζει την κυβέρνηση να φροντίσει για τη δικαιοσύνη. Είδαμε τις φωτογραφίες από τις φυλακές κατά την προεκλογική εκστρατεία με βασανιστήρια στις φυλακές, άτομα που έχουν τραυματιστεί σωματικά και ψυχικά και τώρα ζητούν δικαιοσύνη. Το ίδιο συμβαίνει και με τον κόσμο που νιώθει πως ειναι 9-9.500 άνθρωποι των οποίων η ιδιοκτησία βρέθηκε στα χέρια της προηγούμενης κυβέρνησης. Ο κόσμος ζητάει δικαιοσύνη. Ρωτάω λοιπόν, το Κοινοβούλιο τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να βοηθήσει στην ε, αποκατάσταση της δικαιοσύνης υπέρ εκείνων που αδικήθηκαν, χωρίς όμως από την άλλη μεριά να μπει στον πειρασμό να προχωρήσει σε πολιτική βεντέτα. Γιατί αυτό που ακούσαμε και πριν είναι πολύ σημαντικό η συνεργασία να είναι όχι μόνο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στο εσωτερικό ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση για θέματα που έχουν να κάνουν με το εσωτερικό της χώρας. Η Γεωργία λοιπόν προχωράει στο δρόμο της πλήρους δημοκρατίας, προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου. Πρόεδρε, έχω μια ερώτηση ακόμα, προλαβαίνω, για τις σχέσεις με τη Ρωσία. Στην Τυφλίδα είπαμε ότι στηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας. Εγώ προσωπικά και η ομάδα μου στηρίζουμε την αλλαγή στάσης απέναντι στη Ρωσία. Η Ρωσία και η Γεωργία πάντα θα είναι γείτονε χώρες. Δεν υπάρχει αφιβολία γι' αυτό. Συνεπώς, οι σχέσεις πρέπει να εξομαλυνθούν. Εσείς δείχνετε καλή θέληση, ο Πρωθυπουργό, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και το θέμα της οριοθέτησης του διοικητικού ορίου. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό. Η Γεωργία θέλει περισσότερο να συνεργαστεί με την Ρωσία, από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε αυτήν την οριοθέτηση τη διοικητική. Μία ερώτηση με δύο χιλιόμετρα όμως. Ε. Η κυρία Νέιτς έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, Μαζί με τον συνάδελφο Λίζεκ ήμουν μέλος μιας αντιπροσωπείας η οποία πολύ πρόσφατα επισκέφθηκε την Γεωργία, κύριε πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Γνωριζόμαστε εδώ και κάποια χρόνια και ήταν μεγάλη χαρά και τιμή μου που σας καλωσόρισα και εσάς και το κόμμα σας στους κόλπους της πολιτικής μας οικογένειας με διάφορες ιδιότητες και να σας δώσω οποιαδήποτε υποστηρίξη καταφέραμε να σας δώσουμε με την παρόντα του χρόνου. Είναι μεγάλη μας χαρά λοιπόν που σήμερα σας βλέπουμε στην παρούσα θέση σας και που στη θέση σας αυτή κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να διασφαλίσετε την εύρυθμη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Που έχει περάσει μία συνταρακτική περίοδο συγκρούσεων μεταξύ των διαφόρων πολιτικών δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας πριν από δύο εβδομάδες ε, συναντηθήκαμε με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, της σημερινής αντιπολίτευσης, της ε, μέχρι πρόσφατης ηγεσία και με τους εκπρόσωπους της άλλης πλευράς και πραγματικά είδαμε τις εντάσεις που υφίστανται Καταφέραμε επίσης να μετρήσουμε και μια ορισμένη προθυμία να υπερβληθούν αυτές οι εντάσεις, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στη Γεωργία να προετοιμαστεί για το μέλλον. Του των λεχθέντων, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορώ να αναιρέσω το γεγονός ότι μου προκαλεί αμηχανία το γεγονός ότι παρακολουθώ την πρόσφατη φυλάκιση των πρώην πολιτικών ηγετών. Ασφαλώς δεν είμαστε εμείς εκείνοι που θα κρίνουμε κατά πόσον υπάρχουν ε, πραγματικά λόγοι για τη σύλληψη αυτή, κατά πόσον έχουν διαπραχθεί εγκλήματα. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η υποψία, πλανάται μία υποψία εκδίκησης σε ένα βαθμό στα γεγονότα αυτά αποτελεί κάθε αυτό μία αιτία αμηχανίας, μία αιτία που μας οδηγεί να ζητήσουμε εξηγήσει. Ελπίζουμε, ελπίζουμε στις απαντήσεις σας να είσαστε σε θέση να μας διαβεβαιώσετε ότι οι προσπάθειες μεταρρύθμισης του δικαστικού σώματος θα αφορούν και τον κώδικα ερευνών τον κώδικα για την εξαγωγή των, ε, της δίκαιας δίκης. Ελπίζω να μπορείτε να μας καθησυχάσετε με τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρω ότι μα μας πιέζει ο χρόνος. Πλησιάζει και η συνέδρια κορυφή στην έτσι λοιπόν δεν έχω χρόνο να παραείμε στην διπλωματική πρόεδρε. Δεν είναι ηρωνική η μετάβαση που δηλώσετε ότι έγινε στη Γεωργία γιατί η επιλεκτική δικαιοσύνη εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή σας και αυτό σημαίνει ότι τελειώνει αυτή η ειρηνική μετάβαση. Ακολούθησε ένα επικίνδυνο δρόμο η γεωργιανή κυβέρνηση πολιτικής εκδίκησης και καταστολής της αντιπολίτευσης και αυτό ισχύει για τον πρώην πρόεδρο. Νομίζω ότι ήδη έχετε ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές όπως έγινε και στην περίπτωση της Ουκρανίας και σήμερα λόγω της ε, καταστολής είναι χειρότερη η κατάσταση αν μπορώ να συγκρίνω. Οι δηλώσεις ε, που κάνετε περί ευρωπαϊκής επιλογής ε, και που ακούστηκαν τόσο ωραία δεν είναι πιστευτές αν δούμε τα γεγονότα. Η γεωργιανή κυβέρνηση και το δικαστικό σύστημα παραβιάζει τα ευρωπαϊκά πρότυπα της δημοκρατίας. Δεν ε, πρόκειται για θέμα εδώ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εδώ μιλάμε για την ουσία της δημοκρατίας, γιατί αν φυλακίζετε τους αρχηγούς αντιπολίτευσης, τότε στερείτε το εθνό σας από το δικαίωμα της επιλογής. Θα ήταν καλό αν ε, αληθεύουν ε, οι ευρωπαϊκές σας επιλογές να αλλάξει πρακτική η κυβέρνηση, γιατί αν όχι, η Συμφωνία Σύνδεσης και η Ευρωπαϊκή Προοπτική της χώρας σας θα ξεφοριάσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δεκτεί το δόγμα ε, λιγότερα για περισσότερα, γιατί διαφορετικά θα έπρεπε αυτό να το εφαρμόσει σε όλους τους νότιους και ανατολικούς εταίρους. Ε, εγώ, συζητητής ε, για ε, το θέμα της ανατολικής εταιρικής σχέσης, δεν θα μπορέσω να συστήσω την υπογραφή της συμφωνίας με τη Γεωργία αν δεν αλλάξει η κατάσταση πριν από τη Σύνοδο στο Βίλνιους. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που ήρθατε εδώ. Και εγώ επίσης εκτίμησα το ότι η Υπουργός Εξωτερικών σας ε, τήρησε μια πολύ ειλικρινή στάση στις συνομιλίες που είχε με πολλούς από εμά. Ε, σε σχέση με όσο είπαν ε, και συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να σας ρωτήσω πού βλέπετε ότι οι προσπαθίες σας βελτίωσης, ε, εξομάλυνσης των σχέσεων σας με τη Ρωσία κάπως ουσιαστικά εφαρμόζονται και από την άλλη πλευρά και κυρίως σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική κατοχή. Επίσης, να σας ρωτήσω, αναφερθήκατε σε επεισόδιο, που δεν είναι απλώς επεισόδιο, απλά συνεχιζόταν για πάρα πολλά χρόνια, για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων και αυτό γινόταν ε, με στόχο να εκβιαστούν κάποιοι άνθρωποι. Και φαίνεται να υπονοήσατε πως ε, είχε εμπλακεί ο πρώην Υπουργό Εσωτερικών. Όμως ε, αυτό είναι κάτι που φτάνει μόνο μέχρι τον Υπουργό Εσωτερικών ή υπάρχει και κάποια σύνδεση και με άλλους ανθρώπους ε, από τον κύκλο του Πρωθυπουργού και για ποιο λόγο μπήκε στη φυλακή ο Πρωθυπουργός Ποιες ε, είναι οι ποινικέ κατηγορίες ε, κατά του Πρωθυπουργού αν υπάρχουν ή είναι θέμα πολιτικής βεντέτας, επιλεκτικής δικαιοσύνης όπως υπόθηκε. Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Είπατε ότι το θέμα, συγγνώμη, το σύστημά σας για τις θεωρήσεις ήταν υπερβολικά φιλελεύθερο και φαντάζομαι ότι ίσως ε, αυτό συνδέεται με το ρόλο που έπαιξε η χώρα σας στις σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά στην ευρύτερη περιοχή. Προσπαθείτε να το καταπολεμήσετε. Αυτό είναι προτεραιότητα στρατηγική σας για μια ιστορική μεταρρύθμιση στο θέμα αυτό. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω τον ε, Πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Εγώ ανησύχησα που ε, περιγράψετε τον εαυτό σας ως εκπρόσωπο της ε, γεωργιανής κυβέρνησης. Ε, σίγουρα ο πρόεδρος ε, του Κοινοβουλίου εκπροσωπεί τα συμφέροντα του Κοινοβουλίου του σε ό,τι αφορά και τα δικαιώματα ελέγχου και όχι της εκτελεστικής εξουσίας. Ίσως να υπήρχε γλωσσικό πρόβλημα. Όμως εγώ νομίζω το ίδιο εκπροσωπείται το Κοινοβουλίο σας και όχι την κυβέρνησή σας. Θα ήθελα βέβαια να καλωσορίσω το γεγονό ότι το Γεωργιανό όνειρο δεν έχει τροποποιήσει την πολιτική που κληρονόμησε από την προηγούμενη κυβέρνηση και ιδίω την επιθυμία για καλύτερες σχέσεις με τη Μόσχα. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει ξεπούλημα ε, σε σχέση με το θέμα της κατοχής της επικρατείας σας. Και η δική μου ομάδα έχει σχέσεις όντως με το συντηρητικό κόμμα Τη Γεωργία που ανήκει στο συνασπισμό. Τώρα, εδώ, εκπροσωπώντα όχι την κυβέρνηση, αλλά τον εαυτό σα ω μέλο του κοινοβουλίου σα για το θέμα του Νότιου Καυκάσου και της, ε, το θέμα τη γειτονία. Καλύτερε σχέσει με τη Μόσχα σημαίνει και καλύτερε ε, σχέσει με την Αρμενία. Εγώ είμαι καλό φίλο τη Αρμενία και ε, για καιρό τώρα ε, βρίσκεται κάπως πιεσμένη μεταξύ τη δική σας χώρα και του Ζερμπαϊτζάν και το δικό σας ε, κόμμα Ποια είναι η στάση που τηρεί απέναντι στο στενό συμμαχό του την Τουρκία, δηλαδή ε, πώς ε, βλέπετε και τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Τουρκίας. Eh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε του Κοινοβουλίου που ήρθατε σήμερα εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι συντονιστής εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε αυτή την Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, το ρώτησαν και οι κύριοι Λίσακ και Βόλτσκι για... και είπαν ποια είναι η θέση της ομάδας μας, ότι θεωρούμε ότι είμαστε φίλοι της χώρας σας. Έτσι και εγώ λοιπόν και έχω υποστηρίξει την προσέγγιση της χώρας σας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο στενή συνεργασία δηλαδή ζήτησα, άρα σαφώς και είμαι υπέρ αυτής της συμφωνίας εταιρική σχέσης και συνεργασίας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Αντιλαμβάνεστε τα προβλήματα τα οποία δημιουργούν στην διεθνή κοινότητα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την μετάβαση της χώρας σας. Το κόμμα μου, η ομάδα μου μάλλον, είναι της ίδιας απόχρωσης όπως ε, και ο αρχηγός σας. Θα ήθελα όμως οι δημοκρατικές συνθήκες να είναι οι καλύτερες δυνατόν. Νομίζω λοιπόν πως για μια χώρα η οποία πέρασε από μια διαδικασία επιλεκτικής δικαιοσύνης και βεντέτας, μπορεί να δημιουργούνται παρεξηγήσεις στη διεθνή κοινότητα η οποία να αντιλαμβάνεται τα φαινόμενα αυτά σαν οπισθοχώρηση ή σαν ε, ε, εκδικητική στάση απέναντι σε πολιτικούς αντιπάλους. Εσείς που είσαστε πρόεδρος λοιπόν του Κοινοβουλίου και είσαστε από ένα κόμμα που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό, χωρίς να προκαταλαμβάνουμε βέβαια τα πράγματα, όπως είπε και η κυρία Ακόμες, και χωρίς να λέμε ότι όσοι διώκονται αυτή τη στιγμή είναι αθώοι ή όχι, ρωτάω, τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από τη δικαιοσύνη μήπως θα έπρεπε να είναι λιγότερο δραστικά οι συνθήκες στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Λίσακ μήπως θα έπρεπε να έχουν έτσι ώστε να προστατεύονται περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα των διοκόμενων μήπως θα έπρεπε για παράδειγμα να μπορούν να μένουν υπό περιορισμό σπίτι τους αντί να βρίσκονται στη φυλακή. Η Γεωργία για μας είναι μια χώρα που έκανε βήματα προς τον εξυγχρονισμό. Όλες αυτές οι καταστάσεις λοιπόν βάζουν σε δύσκολη θέση την αξιοπιστία της χώρας σας απέναντι στη διεθνή κοινότητα. Σας το λέω χωρίς να έχουμε ιδεολογικές διαφορές. Απλώς προσπαθώ να καταλάβω, όπως και οι πολίτες που προσπαθούν να καταλάβουν τις αποφάσεις σας σε αυτή την περίοδο μετάβασης που βρίσκεται η χώρα σας. Νομίζω ότι πρέπει να φροντίσετε η δικαιοσύνη να μην αποδίδεται επιλεκτικά και να μην υπάρχουν εκδικητικές στάσεις. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήρθατε εδώ σήμερα. Να ξέρετε ότι εκλαμβάνουμε την παρουσία σας εδώ ως ένα πολύ θετικό σημάδι. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Βάλκ, και εγώ χαιρετίζω την παρουσία σας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω το εξή, έρχομαι από τη Σλοβενία και παραδοσιακά είχαμε πάντα επαφές πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές. Η Γεωργία με τη χώρα μου, την Σλοβενία, ακόμα και παλιότερα, ε, παλιά, όταν η ανεξαρτησία και για σας και για μας ήταν κάτι πολύ μακρινό. Συμφωνώ με τους συναδέλφους εδώ οι οποίοι προειδοποιούν για τις εκδικητικές τάσεις που διαφαίνονται. Αυτοί που φυλακίζονται με πολύ συνοπτικές διαδικασίες, απλώς επειδή συμβολίζουν ή εκπροσωπούν την προηγούμενη κυβέρνηση. Κάνω λοιπόν έκκληση προς εσάς, προς εσάς ο οποίος μου ακούγεστε σαν κάποιος που έχει δημοκρατική στάση. Σας λέω λοιπόν προσοχή. Μερικές φορές δεν ακούγεται καλά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν υποστηρίζουμε τους δικούς μας απέναντι σε άλλους που δεν είναι δικοί μας. Πολύ συχνά, δηλαδή, έχουμε την τάση να μιλάμε με καλά λόγια σε αυτούς που πολιτικά πρόσκειται πιο πολύ σε μας. Όμως υπάρχουν ορισμένες αρχές που είναι πολύ σημαντικές και μία από αυτές είναι ακριβώς να μην εκδικούμαστε. Θέλω να σας ρωτήσω πολύ συγκεκριμένα το εξής. Βλέπετε εσείς παραπάνω δυνατότητες ώστε οι χώρες της περιοχής, όπως η δικιά σας, νομίζετε ότι μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να λυθούν τα προβλήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα ο Καραμπάχ, για παράδειγμα, ή άλλα τα οποία αναφέρθηκαν στις διμερείς σχέσεις. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ θετικό εάν υπάρξουν ιδέες από τη δικιά σας την πλευρά και κάνετε εσείς την προσπάθεια για συνεργασία ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ σας. Εσείς πώς βλέπετε αυτή τη δυνατότητα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας από τη δικιά σας την πλευρά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ για τις τόσο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σας. Σημείωσα όλες τις ερωτήσεις. Φοβάμαι βέβαια ότι δεν θα έχω χρόνο να απαντήσω και σε όλες. Θα κάνω όμως ό,τι μπορώ. Ξεκινώ από το ποιο είμαι, εκπροσωπώ την κυβέρνηση, ποιον εκπροσωπώ. Εκπροσωπώ το συνασπισμό του ονείρου της Γεωργίας και είμαι επικεφαλής. Όλοι στα κόμματά σας έχετε, συμμετέχετε σε συνασπισμούς ή έχετε συνιστώσεις. Εγώ έχω την ευθύνη της πολιτικής ομάδας ως πολιτικός και συγχρόνως Είμαι επικεφαλής στο Κοινοβούλιο. Ως πρόεδρος του Κοινοβουλίου, δεν ξέρω σε τι βαθμό μπορεί ένας τέτοιος πρόεδρος να αναλάβει ευθύνες για αυτά που αποφασίζει το Κοινοβούλιο, πάντως εγώ είμαι επικεφαλής του συνασπισμού το όνειρο της Γεωργίας. Και ήρθα εδώ να σας μιλήσω για τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα μέσα στο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν σας είπα ποιος είμαι και από εκεί και πέρα είμαι έτοιμος να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ρωσία. Νέα πολιτική, κυβέρνηση και τα λοιπά και κατά πόσο οι Ρώσοι κάνουν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Όχι και πολύ. Συμμετέχουν σε συνομιλίες για θέματα Λέγοντα όμω ότι δεν έχει νόημα να μιλήσουν με τον κύριο Σακασβίλη και με την κυβέρνηση. Λέγανε. Τώρα λένε, α, μπορούν να συζητήσουν για κάτι, για κάτι λίγο όμως, με πολύ μικρά αποτελέσματα. Για τα πρώτα φορτηγά με κρασί που μπήκανε στη Ρωσία. Τέτοια μικρά ζητήματα, ναι, αλλά υπάρχει κάτι άλλο. τα προβλήματα που έχουμε με το διοικητικό σύνορο. Έτσι όπως βλέπω εγώ τα πράγματα, το Κρεμλίνο δεν νιώθει καλά όταν η Γεωργία λέει ότι είναι έτοιμη να συζητήσει με συγκεκριμένα θέματα. Προτιμούν να έχουν τα άκρα. Κάποιον δηλαδή ο οποίος λέει όχι σε όλα. Έχει πολύ ριζοσπαστική στάση, δηλαδή κατά. Τότε ξέρουν πώς να τον αντιμετωπίσουν. Ή τους αρέσει και η άλλη άποψη όταν κάποιος λέει ναι σε όλα, ό,τι μου δώσετε εγώ ναι. Ενώ η κυβέρνηση της Γεωργίας είπε και έθεσε τις κόκκινες γραμμές της. Είπε τι δεν είναι διατεθειμένη να δεχτεί. Είπε ότι θέλει την ευρωπαϊκή ε, προσέγγιση κτλ. Είπε τι είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε και τι όχι. Αυτή η στάση δεν κάνει τη Ρωσία να νιώθει καλά και μάλλον σπάει τα νεύρα. Εκείνοι θέλουν ή τη στάση του Σακασβίλη όπως ήταν το 2008 ή τη στάση που έχουν άλλες χώρες στην περιοχή απέναντι στη Ρωσία. Εμείς είμαστε ειλικρινείς και ανοιχτοί και ενημερώνουμε τους Ρώσους και τους λέμε ότι εμείς δεν θα συζητήσουμε ίσα ή μαζί τους. Εκείνοι θέλουν να μειώσουν τη σημασία των συνομιλιών της Γενέβης ή της συνομιλίες που γίνονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούν να έχουν απευθείας επαφές μαζί μας για τα θέματα των συνόρων ή για άλλα, ενώ εμείς τους στέλνουμε το μήνυμα ότι όχι, αυτό δεν θα γίνει. Για το κρασί και για άλλα προϊόντα είναι συζητήσεις για το κρασί και για άλλα προϊόντα. Αν πρόκειται για άλλες συνομιλίες, αυτές γίνονται στη Γενέβη και εμείς δεν θα το αλλάξουμε αυτό. Επί του παρόντος λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν αποτελέσματα. Πιστεύουμε όμως ότι δεν υπάρχει αναλλακτική λύση και κανένας δεν μας έχει προτείνει κάτι διαφορετικό. Είμαστε σε συνεχείς διαβουλεύσεις και επαφές με τους φίλους μας από τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Και οι Ρώσοι το γνωρίζουν αυτό. Ότι δεν υπάρχουν άλλα κανάλια επικοινωνίας μαζί τους. Αυτή είναι η πολιτική μας και θα μείνουμε σε αυτήν. Τώρα, τα μεγάλα θέματα, συγκρούσεις, να πω Καραμπάχ, ε, ε, Σετία κτλ. Η σημερινή Γεωργία δεν νομίζω ότι μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες τώρα. Ίσως ε, με την επανάσταση στο Ρόδο να χάσαμε την ευκαιρία. Μας κόστισε αυτό. Ίσως να μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει τα γεγονότα του 2008. Η καταστροφή αυτή που έγινε στη χώρα θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Και το πήραμε το μάθημα. Έκτοτε αναγνωρίζουμε την πραγματικότητα ότι η Γεωργία δεν μπορεί να αναλάβει τώρα πρωτοβουλίες. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε τη χώρα. Την επικράτεια που είναι υπό έλεγχο δικό μας στη Γεωργία και όχι υποκατοχή. Δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση, αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο έχουμε καταλήξει όλοι, να προτείνουμε κάτι θετικό ούτε για τη διαμάχη στον Αγόρνο Καραμπάχ. Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, Τουρκία, Ρωσία κλπ. Οι γειτονέ μας δηλαδή. οποιοδήποτε παρακολουθεί τα γεγονότα ξέρει πόσο δύσκολο είναι για τη Γεωργία να κρατήσει καλές σχέσεις με όλους. Το προσπαθούμε και το πετυχαίνουμε. Έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Αλλά αυτό απαιτεί καθημερινή προσπάθεια. Με το Αζερμπαϊτζάν σκεφτόμαστε κάποια νέα προγράμματα στο ενεργειακό. Δυστυχώς η Αρμενία δεν συμμετέχει. Η Γεωργία θα ήθελε να είναι το σημείο εκκίνησης και να υπάρξει έτσι ασφάλεια για όλους αλλά δεν γίνεται. Συγχρόνως, ένα πράγμα θα σας αναφέρω. Η προηγούμενη κυβέρνηση αναγνώρισε την γενοκτονία των Τούρκων. Έχουμε την Αρμενία, νότια της χώρας μας. Και για λόγους που αντιλαμβάνονται πολύ καλά οι Αρμένοι, δεν το κάνουμε επειδή είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα, γιατί υπάρχει και η Τουρκία. Αυτό το θέμα της πολιτικής δεν νομίζω ότι βοήθησε. Έδωσε καλά αποτελέσματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και θα είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και τις θεωρήσεις ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Θα υπάρξουν κάποιες υπηρεσίες και στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ως ένα πολιτισμένο σύστημα συλλογής δεδομένων για να διασφαλίσουμε τα σύνορά μας, θα εφαρμόσουμε ό,τι πρέπει να εφαρμόσουμε. Όσον αφορά το έγκλημα, ελπίζω πιστεύω ότι αυτά που γίνονται δεν είναι ευρεία κλίμακος. Ε, σίγουρα πρέπει να προστατεύσουμε καλύτερα τα σύνορα. Αυτό προς πάσα κατεύθυνση. Εννοείται. για την επιλεκτική δικαιοσύνη. Για εννέα χρόνια 99,9% των δημοσίων υπαλλήλων από τα χαμηλά επίπεδα μέχρι τα ψηλά επίπεδα είναι από ένα, ήταν από ένα κόμμα, από το United National Movement. Δεν υπήρχε περιθώριο για κανέναν άλλον, μόνο για ανθρώπους του κόμματος αυτού. Συνεπώς, όλες οι περιπτώσεις, όλα αυτά τα εννέα χρόνια που ερευνώνται μας οδηγούν σε εκπροσώπους του UNM του κόμματος, όχι του Ρεποπλεκανού κόμματος όπου προέρχομαι εγώ, γιατί έτσι κι όλοι οι άλλοι απεκλείονταν. Οπότε δεν εκπλήσει το γεγονός ότι από τις έρευνες καταδεικνύονται οι προσκύμενοι στο UNM, μα δεν υπήρχε και κανένας άλλος. Ποιος ε, παρακολουθούσε τον κόσμο. Σε επίπεδο τοπικής αστυνομίας. Το υλικό φυλάσσεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και δεν το ξέρανε οι ανώτεροι. Χιλιάδες άνθρωποι μας γράφουν και λένε ότι υπογραφή στο χαρτί Α, οι ίδιοι λέγανε ότι χαρίζανε την ιδιοκτησία τους στο κράτος και τώρα το ζητάνε πίσω. Μα ποιος θα μπορούσε να το είχε κάνει αυτό. Ποιος θα μπορούσε να είναι υπεύθυνο για ένα τέτοιο σύστημα. Κάποιοι από εσά ε, έχετε έρθει στην Τυφλίδα. 200 εκατομμύρια μας ε, σύστησε, μας τύχησε η δημιουργία του κέντρου. Από πού έχουν έρθει τα χρήματα, ποιος πλήρωσε τους λογαριασμούς του κτηρίου που φτιάξαμε, που δεν έχει τελειώσει. Τι διαπιστώνουμε. Ότι δεν ήταν από τον προπολογισμό, ότι είχε δημιουργηθεί μια ειδική μονάδα, ότι η κρατική περιουσία δόθηκε στην μονάδα αυτή και ένα εκτάριο της γης ξαφνικά πουλιέται 10 φορές παραπάνω από την τιμή αγοράς εκείνη την περίοδο. Πώς? Να, γιατί ερχόταν ο κόσμος και έλεγε το Υπουργείο Δικαιοσύνης με συμβούλευσε να αγοράσουμε αυτή τη γη γιατί τη χρειαζόταν για να χτίσει εκεί το κτίριο. Και πληρώσαμε 10 φορές παραπάνω, ενώ κανείς δεν χρειαζόταν αυτή τη γη, αυτή την ιδιοκτησία. Αλλά μας ανάγκασαν να το κάνουμε. Τι κάνει λοιπόν κανείς σε αυτές τις περιπτώσεις και πώς αντιμετωπίζει τέτοια ζητήματα. Μαθαίνουμε βέβαια. Γίνανε σφάλματα, αλλά πρέπει να συγχωρηθούν γιατί αλλιώς θα κατηγορηθούμε ότι είμαστε εκδικητικοί. Εντάξει, να παραιτηθούμε από αυτό το πόλεμο. Γι' αυτό και εξάλλου προσφέρουμε αμνηστία στα μέλη της θέως κυβέρνησης, Στην μειοψηφία δηλαδή. Εκεί είμαστε έτοιμοι να δώσουμε αμνηστία σε όλους. Αλλά όχι στους υπουργού και στους παραπάνω, γιατί πρέπει να δώσουμε μια απάντηση στο λόγο της Γεωργίας, γιατί στο κάτω-κάτω σε αυτούς ανήκει η χώρα και είναι θύματα τέτοιων καταστάσεων. Ποια είναι η συμβουλή σας, συγχωρήστε τους όλους ό,τι και αν έχουν κάνει. Ε, ναι, αλλά τότε συμβουλέψτε μας και για κάτι άλλο τότε τι σημαίνει δικαιοσύνη. Πώς θα θέσουμε σε εφαρμογή τη δικαιοσύνη. Ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω εδώ του Μαΐου του 2011 για τη Γεωργία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει από την κυβέρνηση της Γεωργίας να ερευνήσει με διαφάνεια ε, τις ε, υπόνοιες κατά της αστυνομίας. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις. Ελπίζω να παρακολουθήσατε τις εξελίξεις για αυτή την υπόθεση. Στενά. Ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Απρίλιο 2011. Το δικαστήριο εκπλήσεται για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την εξουσία του Υπουργείου Εσωτερικών, ε, η εισαγγελία το τμήμα φυλακών, ο πρόεδρος στο κοινοβούλιο. Σχετικά με επίοικια, ε, για τη δικαιοσύνη όσον αφορά σε περιπτώσεις δολοφονίας. Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν κατά του Μεραμπουσίλη που, ήταν, πριν από τρεις μήνες γενικός ε, γραμματέας, ήταν υπουργό εσωτερικών 8 χρόνια. 8 χρόνια με τον Υπουργό Δικαιοσύνη, τον κύριο Ντιουσφίλη, ο οποίος έφυγε αμέσως μετά τις εκλογές από την χώρα. Να, δύο κέντρα εξουσίας στη Γεωργία Όποιο θέλει να παρακολουθήσει τη Γεωργία πρέπει να το ξέρει αυτό. Αλλιώ πώ το παρακολουθεί. Και ποιε ήταν οι κατηγορίε. Μακάρι, πώ να το πω, να μην ήμουν υποχρεωμένο να σα τα πω αυτά. Γιατί πολλέ φορέ σα έχουμε πει στείλτε παρατηρητέ. κύριο Χάμερβερτ. Δύο εβδομάδες ήταν στη Γεωργία, δύο εβδομάδε εδώ και έχει πρόσβαση σε όλο το υλικό, σε όλες τις ε, δικαστικές ακροάσεις. Και εμείς θέλουμε και άλλους παρατηρητές. Γιατί αυτά που σας λέω εγώ, το καταλαβαίνω, είναι λόγια που σας λέω εγώ. Δεν μπορείτε να με θεωρήσετε ότι μεροληπτώ. Αλλά ο κύριος Μεραποσβίλη, γιατί κατηγορείτε. Τον Ιούλιο έγινε, στις 4 Ιουλίου έγινε υπουργό. Στις 15 Ιουλίου δύο υπουργοί υγείας και κοινωνικής προστασίας, 22 άτομα προσελήφθησαν. 22.000, ναι. Τρεις μήνες πριν από τις εκλογές. Γιατί? Για να μετράνε τους άνεργους στη Γεωργία. Έρχεται λοιπόν με αυτή την πρόταση. 1η Οκτωβρίου έχουμε εκλογές και το Σεπτέμβριο 22.000 Γεωργιανοί προσλαμβάνονται, πληρώνονται από το κράτος για να μετράνε τους άνεργους. Και αυτοί 22.000 λένε τι κάνανε αυτό το μήνα το Σεπτέμβριο που δουλεύανε. Χρησιμοποιήθηκαν στο κόμμα, το UNM, ένα μήνα πριν τις εκλογές. Ναι. Και πάλι, όπως σας είπα και πριν, θα προτιμούσα να μην χρειαζόταν να σας πω τέτοια πράγματα, να σας τα πω αυτά. Αλλά γι' αυτό κάνω έκκληση. Μην πιστέψτε εμένα. Αλλά μην πιστέψτε άλλους που πολιτικά μεροληπτούν αυτούς που είναι μόνο στην κυβέρνηση. Όχι. Πιστέψτε το Human Rights Watch, τη Διεθνή Αμνηστία, τους ανεξάρτητους. Τέλος, σχετικά με αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις που μου υποβάλλατε και τις συστάσεις σας και να ξέρετε ότι τα παίρνω όλα πάρα πολύ σοβαρά. Και είμαι έτοιμος να συνεχίσω. Συγχρόνως όμως, επιστρέφοντας, παίρνω ένα δίδαγμα από τη σημερινή συζήτηση. Και αυτό είναι το τι είναι επιλεκτική δικαιοσύνη. Κύριε Βόλσκι, μου δίνετε ένα καλό μάθημα. Τι είναι επιλεκτική πολιτική δικαιοσύνη. Όταν ξέρουμε τι θέλουμε και το λέμε. Γιατί η επιλεκτική πολιτική δικαιοσύνη μπορεί να λάβει χώρα όχι μόνο στη Γεωργία, αλλά και αλλού αν λοιπόν ήδη ξέρετε ότι έτσι έχουν τα πράγματα στη Γεωργία, τότε η Γεωργία δεν πρέπει να πάρει τίποτα παραπάνω. Το δηλώνεται. Ένα. Ε, αυτό είναι. Επιλεκτική πολιτική δικαιοσύνη, που εγώ δεν πρέπει να το κάνω. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Σας ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Έχετε λίγα δευτερόλεπτα κύριε Πρόεδρε. Και αυτό σα εμπλέκει στο ρόλο σα ω Πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Μιλήσατε για τη νέα έδρα του Κοινοβουλίου και τώρα τις ε, κατηγορίες ε, για την ενώθευση των τιμών ε, τη γη κτλ. και ενδεχόμενη διαφθορά σας. Ρωτώ γιατί είμαι κατά του Στρασβούργου και τη έδρα του Στρασβούργου και το τσίρκο και τα χρήματα που ξοδεύονται. Η κυβέρνησή σα, ο κυβερνητικό σχηματισμό εξετάζει να επιστραφεί το κοινοβούλιο στην Τυφλίδα και να σωθούν αυτά τα χρήματα, να εξοικονομηθούν αυτά τα χρήματα που επιβαρύνουν τον προλογούμενο αυτή τη στιγμή στη Γεωργία. Αν ναι, παρακαλώ να το δηλώσετε. Okay. Uh, the answer, the answer. Η απάντηση on, on, on the parliament, first of all. για το θέμα του Κοινοβουλίου καταρχάς. Θέλουμε να έχουμε όσο πιο στενέ σχέσει γίνεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε όλου όσου ε, ε, επισκέφθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το παλιό κοινοβούλιο μα, Θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τα διοκτήρια και τα χρήματα του φορολογούμενου. Έγιναν αλλαγέ και τροποποιήσει του Σύνταγμα που ε, επιτρέπουν να λειτουργήσει το Κοινοβούλιο και στην Τυφλίδα προκειμένου να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να είμαστε πιο κοντά στην πολιτική ζωή, στα πολιτικά τεκτενόμενα, το οποίο δεν συμβαίνει σήμερα και σε πολλές περιπτώσεις όταν ο κόσμος επισκέπτεται τη γεωργία δεν είμαστε σε θέση να συναντηθούμε γιατί δεν βρισκόμαστε εκεί και με τους εμπλεκόμενους φορείς του Κοινοβουλίου οι οποίοι είναι μακριά. Προσπαθούμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε με καλύτερο τρόπο τα χρήματα του φορολογούμενου και τα χρήματα τα οποία δαπανώνται ακόμα και σήμερα για την ε, διοργάνωση εκδηλώσεων κτλ. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρήματα του προλογούμενου, το δημόσιο χρήμα αλλά και το ιδιωτικό χρήμα, γιατί δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να φορολογούνται οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με σωστό τρόπο τα χρήματα αυτά. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Σάριος Βόλφσκι ήθελε να θέσει μία ερώτηση ακόμα, αλλά αν ξαναξεκινήσει η συζήτηση δεν θα έχουμε χρόνο να περάσουμε στα επόμενα θέματα. Δεν θα ξαναρχίσω. Μας είπε ο κύριος Κασμεσφίλη ότι θα βάλουμε τον κόσμο στη φυλακή για να δώσει υποδειγματικό, με υποδειγματικό τρόπο τι θα γίνει με αυτούς που είναι αντίθετο. Το είπε αυτό στην κυρία Φρατίνη. Απάντηση. Να σας πω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Δεν στέκει αυτό. ότι θα μάθει, θα προσπαθήσει να δώσει ένα μάθημα σε όσους είναι αντίθετοι σε αυτόν. Αυτή είναι η κατηγορία. Αλλά αυτό να μου το επιβεβαιώσει όποιος ήταν στην συνάντηση εκείνη. Ο, αν είπε ο Πρωθυπουργό ότι θα τιμωρήσει όποιον ε, του αντιταχθεί. Ο κ. Σακασβίλης το έκανε αυτό. Ο κ. Σακασβίλης το έκανε αυτό. Και παρακαλώ να δω τα πρακτικά της συνάντηση ή να δω κάποιον ο οποίο να ήταν στη συνάντηση εκείνη με τον Πρωθυπουργό. Τι λέτε. Μάλιστα λέει ο πρόεδρο. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σα ευχαριστούμε που ήρθατε στην Επιτροπή μα που απαντήσατε τι ερωτήσει μα. Δεν είναι πάντα ευγενικέ οι ερωτήσεις, αλλά νομίζω ότι ο διάλογο θα πρέπει να συνεχιστεί. Σα ευχαριστώ εγώ πολύ και προσβλέπω στην μελλοντική συνεργασία και από πλευράς ε, και εδώ πέρα και στην Γεωργία.